Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ πολύ. Όταν ολοκληρωθεί και η συζήτηση ανάμεσα στο ΕΛΚ και τους σοσιαλιστές, Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Δευτέρα, νωρί το απόγευμα. Ξέρω ότι η Δευτέρα είναι προβληματική μέρα για πολλούς συναδέλφους. Ξέρετε πάντως ότι είναι μια εβδομάδα συνεδρίασης πολιτικών ομάδων. Πολλές αίθουσες την Τρίτη και την Τετάρτη είναι κατελημένες από τις συνεδριάσεις των πολιτικών ομάδων και έτσι κι εμείς όπως και άλλες επιτροπές αναγκαζόμαστε ουσιαστικά να συνεδριάσουμε ιδίω για τις ψηφοφορίες τη Δευτέρα το απόγευμα. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Η ψηφοφορία για την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το σημείο 7 δηλαδή της ημερήσιας διάταξης, αναβάλλεται για τον Ιανουάριο. Το σημείο 10, Προπολογισμό 2017 όπου εξετάζουμε αιτήσει μεταφοράς, θα το εξετάσουμε μετά το σημείο 4, όπου θα ασχοληθούμε με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και πριν από τις προφορίες που θα ξεκινήσουν στις 4 ε, παρατέταρτο. Δεν υπάρχουν κρεμμοί ε, εκκρεμεί αιτήματα μεταφορών για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τον κύριο Γκέιερ, λοιπόν, θα δούμε τι έχει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τον κύριο Ρέλ μαζί μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία του, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την εκτέλεση του προπολογισμού, ιδίως όσον αφορά τα αυτόνομα εμβάσματα, τα οποία έγιναν πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα το σημείο 13, κτηριακή πολιτική, ενημέρωση προκατακτική μάλλον ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης αναβάλλεται και αυτό, γιατί δεν έχουμε εδώ πέρα την συγκεκριά μας την κυρία Μόνικα Χολμάιερ. Έχετε λάβει τα συμπεράσματα των, της συνεδρίσεως των ιστών της 23ης Νοεμβρίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι εγκρίνονται οι αποφάσεις αυτές οριστικά πλέον. Και σας προτείνω να μου πείτε αν υπάρχει κάποια αντίρρηση για τα σχέδια πρακτικών της 10ης-11ης 11 η 14ης η 9ης 10ης Οκτωβρίου, 9ης η νοεμβριου 22ης-23ης Νοεμβρίου. η νοεμβριου λάβει γνώση των συμπερασμάτων αυτών. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Μπορούμε να εγκρίνουμε λοιπόν τα σχέδια πρακτικών. Να σας παρουσιάσω τώρα τη δική μου τη γνωμοδότηση όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ασχολούμεθα με ένα ζήτημα το οποίο μας έχει απασχολήσει προφανώς και στο παρελθόν. Ξέρετε ότι ζητήσαμε μία μελέτη από εξωτερικούς πυρογνώμονε όσον αφορά την αναγκαιότητα να συντονιστούμε καλύτερα και να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο συντονισμό και με καλύτερη συνέργεια ανάμεσα σε ευρωπαϊκές και εθνικές δημοσιονομικές πρακτικές προκειμένου να έχουμε τις καλύτερες δυνατές επιπτώσεις όσον αφορά την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη. Στο σχέδιο λοιπόν έκθεση, στο σχέδιο γνωμοδότησης το οποίο σας υποβάλλω, το οποίο είναι ιδιαίτερα λακωνικό όπως βλέπετε, έχει μόνο πέντε σημεία, επιμένω στο ζήτημα αυτό, της αναγκαιότητας αυτού του συντονισμού και λέω ότι στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να μας απασχολήσει το συνολικό αυτός, ιδίως όσον αφορά την περίοδο μετά το 2020. Νομίζω ότι όντως θα πρέπει να επιτευχθούν οι απαραίτητες συνέργειες ανάμεσα στους εθνικούς προπολογισμούς και στον κοινοτικό προπολογισμό. Και δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια άμεση διασύνδεση ανάμεσα στα δύο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να φέρει πέρα όλες τις μεταρρυθμίσεις που έχει ξεκινήσει και θα πρέπει να κάνει και μία παρουσίαση πλέον, μία ανακοίνωση όσον αφορά τους νέους ιδίους πόρους. Ο κύριος Λεβαντόφσκι και ο κύριος Ντεμπρέ θα μας κάνουν μία ανακοίνωση προς αυτό σε λιγάκι και περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε τι θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της δέσμης μέτρων προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε μια δημοσιονομική αν μη τι άλλο ικανότητα της Ευρωζώνης προκειμένου να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τους συμμετρικούς ή ασυμμετρικούς κλειδονισμούς και να καταφέρουμε τελικά να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουν να ολοκληρώσουν τις μεταρρυθμίσεις τους, να έχουν τα απαραίτητα μέσα στα πλαίσια ενός συστήματος προϋποθέσεων και ρεσιμότητος. Με ικανοποίηση επίση μπορούμε να χαιρετήσουμε την πρωτοβουλία που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον μετασχηματισμό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που θα πρέπει να πάρει τη μορφή ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου για την Ευρωζώνη. Αυτά λέω πάνω κάτω στο σχέδιο αυτογνωμοδότησης. Αυτά θεώρησα ότι θα πρέπει να τονιστούν σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο βάσει του άρθρου 54. Ξέρετε ότι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων. Οι συνάδελφοι και οδησηγητές μπορούν να πάρουν τώρα το λόγο. Ιβάν Στέφανε πρώτος. Είναι παρόν. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για το γεγονό που ανέφερε στα βασικά σημεία σχετικά με αυτό το φάκελο. Εγώ θα επανέλθω στα θέματα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό, παραδείγματο χάρη, ο συντονισμό, η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ όλων των ε, οικονομικών πολιτικών των χωρών ε, της Ευρωζώνης αλλά και σε ό,τι αφορά τη μετατροπή ε, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Ε, πρέπει να μιλήσουμε για του ιδίου πόρου βέβαια και αυτά που είπατε είναι ακριβώ αυτά που στηρίζουμε και εμεί. Από εκεί και πέρα θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Ο σημείο 6 έχει να κάνει με τις ε, χώρες που δεν έχουν ακόμα προσχωρήσει στο ευρώ δεν έχουν ακόμα το ευρώ ως μονάδα, αλλά πρέπει να προετοιμάσουν το σχέδιο δράσης τους για να εφαρμόσουν ε, το σχέδιο αυτό, διότι όσοι ε, δεν έχουν ακόμα ευρώ, αλλά έχουν συμφωνήσει να, το, να προσχωρήσουν σε αυτό κάποια στιγμή, ε, θα πρέπει ε, να τους ενθαρρύνουμε ότι θα ακολουθούν μια πολιτική ευθυγραμμισμένη με τη δική μας Ευχαριστώ. Ναι, βεβαίως το ευρώ είναι το νόμισμά μας και όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κάποια στιγμή ε, θα προσχωρήσουν στην Ευρωζώνη, εφόσον το επιθυμούν βέβαια και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Ο συνάδελφος Ντοσάντος. Εκτός μικροφώνου όμως ο κύριος Ντοσάντος δεν τον ακούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που υποβάλλετε αυτή η γνωμοδότηση. νομίζω ότι συνοψίζει τα κεντρικά ζητήματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές μας τουλάχιστον για το συγκεκριμένο φάκελο. Δεν είμαστε εμείς η αρμόδια επιτροπή κατά κατά κύριο λόγο. Ε, ήταν πολύ σωστά πάντως που είπατε, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής. Ε, θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για το έγγραφο. Επίσης, αυτά τα έγγραφα είναι πάντα σύντομα. και μου έκανε εντύπωση που μπορέσατε εσείς αυτόν το συνοψίσετε σε πέντε προτάσεις που είναι οι βασικές πτυχές του ζητήματος. Για να δούμε και πώς η, Επιτροπή, η Δημοσιονομική Επιτροπή μπορεί να συνεισφέρει και αυτή ε, στο ζήτημα αυτό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Βεβαίως υπάρχει το θέμα των εθνικών προπολογισμών, υπάρχει το θέμα του ευρωπαϊκού προπολογισμού και το θέμα των ιδιών πόρων. Επίσης η αιτήσια με έρευνα ανάπτυξης και αυτή είναι σημαντική. Είναι σημαντικό όλα αυτά τα στοιχεία τα κράτη-μέλη να τα ε, εντάξουν στις οικονομικές τους πολιτικές. και βεβαίω ε, λαμβάνεται υπόψη και ο μηχανισμό ε, το σύμφωνο σταθερότητα. θέλουμε να έχουμε μια σημαντική δυνατότητα σε επίπεδο ευρωπαϊκού προπολογισμού που να χρηματοδοτείται από του δύο σπόρου. Και αυτό είναι καλοδεχούμενο στην πρότασή σα. Δεν είναι εύκολο βέβαια, αλλά σιγά σιγά βλέπουμε φως στο βάθος του τούνελ, όλο και πιο πολλά κράτη-μέλη, όλο και πιο πολλοί πολιτικοί θυνούντες αντιλαμβάνονται ότι είναι κάτι επί το οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε. Το κοινό ευρωπαϊκό μας σχέδιο περνάει από μια καλύτερη κατανομή των δυνατοτήτων, των πόρων από ό,τι μέχρι τώρα. Επίσης συμφωνώ με τον προηγούμενο ομιλητή όταν λέει ότι θα πρέπει να αναφερθούμε και στις χώρες που προετοιμάζονται ε, για να ε, ενταχθούν στην Ευρωζώνη. Συμφωνώ δηλαδή με τις ανησυχίες του συναδέλφου. Το είπε και ο Επίτροπος πρόσφατα. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό το θέμα να συμπεριληφθεί στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριος Κόλμπελ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρα. Και καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά που κάνατε μαζί με τον συνεισήγητη. Ωστόσο, κάπως έχω ενοχληθεί σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις αυτές και ιδιαίτερα όταν ακούω ότι το ευρώ το χαρακτηρίζουμε ως μια επιτυχή ιστορία. Μα που ζούμε. Το ευρώ αποτελεί μια ιστορία μία σύμβαση ε, η οποία έχει ήδη παραβιαστεί εκατοντάδες φορές. Εξακολουθεί να εμφίσταται το ευρώ σήμερα γιατί ε, χρησιμοποιούνται πακέτα διάσωσης διαρκώς και αφότου ούτε αυτά δεν ε, άρκεσαν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε αντίθετα με τις ανάγκες της αγοράς να μηδενίσει τα επιτόκια και να εισαγάγει και ένα σύστημα ομολόγων το οποίο θεωρούμε ότι είναι σαφής παραβίαση της εντολής της ΕΚΤ. Πρόκειται για παραβίαση του δικαίου και το ότι το χαρακτηρίζουμε αυτό ως ιστορία επιτυχίας πραγματικά με αφήνει έκθαμβο. Σε ό,τι αφορά το ευρώ, θεωρώ ότι θα πρέπει να δηλώσουμε τις ε, προθέσεις μας. Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε μόνο τα όσα συμβαίνουν. Θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους, γιατί το ευρώ δεν μπορούμε να το συντηρήσουμε τεχνητά διαρκώς με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέχρι ότου φτάσουμε σε υποπληθωρισμό. Αν θέλουμε και αν έπρεπε να υπάρχει ένα κοινό ενιαίο νόμισμα, θα έπρεπε να αναγνωρίζουμε και τα προβλήματα τα οποία είναι εξή, ότι έχουμε ομαδοποιήσει χώρες οι οποίες από πλευράς οικονομικής απόδοσης δεν ταιριάζουν μαζί. Δεν είναι αυτό, προφανώς είναι κρίμα για τις χώρες αυτές που έχουν χαμηλότερη απόδοση, αλλά πολύ απλά θα πρέπει να το ομολογήσουμε. Αυτό που είναι πραγματικά κατακριτέο είναι ότι προσπαθούμε να συντηρήσουμε ένα νόμισμα το οποίο ε, δεν είναι συντηρείται από μόνο του και θα διχάσει την Ευρώπη. Και πραγματικά θα ήθελα να μας προειδοποιήσει όλους μας να μην συνεχίσουμε στον δρόμο αυτό. Ευχαριστώ για αυτή την ε, σταθερότητα στην ανάλυση, τη συνέπεια. Άλλος κανείς, ο κύριος Ντεναντό έχει το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, ακούστε, αν θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι οικονομικό επίπεδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να έχουμε και τα κατάλληλα μέσα. Και αυτό σημαίνει να επιλύσουμε επιτέλους το θέμα των ιδίων πόρων. Να υπάρχει ένας προϋπολογισμός ε, ε πραγματικός για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Χαίρομαι που κάνατε αυτή την ανάλυση. Ε, από εκεί πέρα βεβαίως θα πρέπει η Ευρωζώνη ε, να εδραιωθεί. Εγώ πιστεύω πως είναι ε, πλούτος για την Ευρώπη. να με τον προηγούμενο μιλητή η Ευρωζώνη. Τώρα που φεύγει το Μένο Βασίλειο υπάρχει χώρος για, ε, για άλλα για να ε, ενταχθούν στην Ευρωζώνη. Θα πρέπει να διβερθεί η Ευρωζώνη, αλλά βεβαίως δεν πρέπει να τρομάζουμε τους υποψηφίους. Νομίζω ότι έχουμε κάθε συμφέρον όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να προσχωρήσουν στην Ευρωζώνη γιατί είναι, επαναλαμβάνω, η κοινή μας περιουσία. Βρισκόμαστε σε μια καμπή αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ε, όπως το παρελθόν. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτόν τον ε, προϋπολογισμό τον ισχνό. Χρειαζόμαστε να έχουμε τα μέσα για να μπορέσουμε να ασκήσουμε την πολιτική που θέλουμε. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ούτε εγώ συμφωνώ με τον κύριο Κόλμερ αυτός λέει ότι το ευρώ δεν πέτυχε. Εγώ λέω το αντίθετο. Το ευρώ έδειξε την ισχύ της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Επίσης, βεβαίως, έδειξε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ε, αυτή η οικοδόμηση της Ευρωζώνης. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, τους κατάλληλους μηχανισμούς για να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Πάντως σίγουρα η κρίση δεν ευθύνει, για την κρίση δεν ευθύνεται το ευρώ ε, και πολλές χώρες μάλιστα σώθηκαν επειδή συμμετείχαν στην Ευρωζώνη και είχαν την κατάλληλη υποστήριξη. Εν πάση δεν ζήτησα το λόγο γι' αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν συνδέεται βέβαιω άμεσα με τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, αλλά μεταφράζεται και στο δημοσιονομικό επίπεδο και είναι το κοινωνικό σκέλος. Διότι όταν μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, μιλάμε για μακροοικονομικά μέτρα, μιλάμε για κάποια αριθμητικά στοιχεία ε, μεγάλης κλίμακας, αλλά δεν δίνεται αρκετή έμφαση στην, στον, στον κοινωνικό πυλώνα, στην κοινωνική πολιτική. Πριν από, μία, πριν από λίγες εβδομάδες στον Κέντεμπορκ επιτέλους ε, υπεγράφει μια πριν απο λιγες αυτό στον κεντεμπορκ επιτελους υπεγραφει μια συμφωνια για αυτό τον κοινωνικό πυλώνα, ε, θα ήταν καλό λοιπόν αυτές τις, αυτές τις συστάσεις ε, να περιλαμβάνουν και, και το κοινωνικό σκέλος. Δεν συνδέεται άμεσα με τον προπολογισμό βέβαια αυτό, αλλά ε, συνδέεται με το πώς θα, θα συνδυάσουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό με το ευρωπαϊκό εξάμεινο. θα πρέπει λοιπόν και το κοινωνικό σκέλος να αναφέρεται και εδώ στην, Επιτροπή, στην Δημοσιονομική Επιτροπή. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Όβαρτ. Um, uh, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την δουλειά που έχετε κάνει. Για το θέμα του ευρώ. Έχουμε διάφορους προφήτες τέτοιων καταστροφών στο Ενωμένο Βασίλειο που προέβλεπαν την κατάρρευση του νομίσματος από την ίδρυσή του. Και αυτό ακόμα δεν έχει συμβεί. Και ούτε Πρόκειται για την μεγαλύτερη οικονομική κρίση λόγω του ευρώ των τελευταίων 100 χρόνων και νομίζω ότι λίγο πίστη παραπάνω και λίγο πιο επικοδημητικό πνεύμα δεν θα έβλαπταν. Εγώ σίγουρα δεν βλέπω να καταραίει όπου να είναι το ευρώ. Σε ό,τι αφορά τώρα την γνωμοδότηση κάθε Νομίζω ότι τα στοιχεία είναι εντάξει, αλλά ίσως σε κάποια φάση θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κάποιες ρήτρε για τη γενική κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την ε, χρηματοδότηση, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, την καινοτομία, τις μικρομεσαίες. Γιατί όπως σας είπαμε, συζητήσαμε το τελευταίο καιρό τόσο εμπισταμένο στον προπολογισμό του 2018 σε θεωρητικό επίπεδο. Μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις στον κλάδο της απασχόλησης, στην ανάγκη συμπερίληψη πρωτοβουλειών και στην πρωτοβουλία για τους νέους και επίσης να τονίσουμε την ανάγκη για δίκαιη φορολόγηση σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε παρατηρήσεις για την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το θέμα των φορολογικών παραδείσων, των ε, εταιριών offshore, των ε, εταιριών, των κούφιων εταιριών σε ό,τι αφορά την ε, αποφύγη κατά φόρων, σε ό,τι αφορά τέτοια έσοδα για τον ευρωπαϊκό προλογισμό, προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερου πόρου για να επενδύσουμε στου τομεί που μα ενδιαφέρουν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριος Φερνάντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι περίεργος ε, για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια νέα γραμμή του προϋπολογισμού μέσα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια γραμμή για την ενίσχυση της Ευρωζώνης ως, ε, αν θέλετε, μια ενδιάμεση στάση προς μια τραπεζική ένωση. σε ό,τι αφορά και την αντιστάθμιση ασύμετρων κλειδονισμών. Δεν θα βοηθήσει απλά τα κράτη-μέλη στην Ευρωζώνη, αλλά και αυτούς που προτίθενται να μπουν στην Ευρωζώνη. Και τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις ε, που είναι απαραίτητες. Είμαι περίεργος λοιπόν να δω πώς ε, θα πώς οι πόροι θα δαπανηθούν στη γραμμή αυτού του προπολογισμού και αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι πολύ ευτραφής προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά το 1% του Εθνικού ΕΠ. Ελπίζω αυτή η γραμμή του προπολογισμού, την οποία και υποστηρίζω, να μην καταλήξει, να μειώσει τον προπολογισμό τη Ευρωζώνης. Ελπίζω να μπει επιπροσθέτω, όπως και θα έπρεπε άλλωστε. Επίσης, ζητούμε πολλά από τον Ευρωπαϊκό προπολογισμό και σε κάποιε περιπτώσει. Ε, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί, όχι λόγω όγκου, αλλά και γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχουμε αρμοδιότητες σε οικονομικά, φορολογικά θέματα, θέματα εκπαίδευσης. Αυτές είναι αρμοδιότητες ε, των κρατών μελών. Εμείς μόνο ε, είμαστε, υποστηρικτικά λειτουργούμε. 60% των δημοσίων ταπανών στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, προέρχεται από κοινωτικούς προϋπολογισμούς, από κοινωτικό προϋπολογισμό. Και αυτό καταδεικνύει ότι όσο μικρός και αν είναι αυτός ο προπολογισμό, συνεισφέρει τα μάλα στα κρατημέλη. Και το 2018 έχουμε ένα στόχο για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Καταφέραμε να βρούμε μια καλή συμφωνία και είμαι πεπισμένο ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα βοηθήσει στην ανταγωνιστικότητα, στη συγκοινωνική συμπερίληψη και επίσης ε, θα συμβάλλει και στην ασφάλεια την οποία χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντό των ορίων που ανέφερα λοιπόν, φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη έχουν ακόμα αρμοδότητε. Δεν νομίζω ότι θέλει να πάρει κανεί άλλο το λόγο. Α ολοκληρώσουμε λοιπόν τη συζήτηση. Νομίζω ότι το ευρώ ανταποκρίθηκε ουσιαστικά στην αρχική αποστολή του όποια και αν είναι άποψή μας κύριε Κόρμελ. Γιατί ξέρετε ότι έχουμε πλέον μία ενιαία αγορά και είχαμε στο παρελθόν ξεχωριστό νόμισμα για κάθε χώρα. Στα τέλη λοιπόν της δεκαετίας του 90 η συναγματική ισοτιμία, η σταθερότητα της συναγματική ισοτιμία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς γινόταν πλέον ένας παράγοντας μείωσης οικονομικής ανάπτυξης και ακόμα και ανεργίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύ μεγάλη αστάθεια και προκειμένου να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες σταθερότητας χρησιμοποιήσαμε την, το νέο νόμισμα. Δεν ξέραμε αν έπρεπε να υπάρχει εκείνη τη στιγμή μια κοινή οικονομική, ε, νομισματική ε, διακυβέρνηση. Υπήρχαν ορισμένες χώρες τότε, οι οποίες ε, αντιτάχθηκαν στην ιδέα αυτή μιας οικονομικής, νομισματικής, δημοσιονομικής διακυβέρνησης. Και για αυτό το λόγο δημιουργήσαμε το καθεστώς αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα, το Eurogroup. Το Eurogroup βέβαια δεν κυβερνούσε εντό αγωγικών. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επέβαλε κυρώσει στι παραβάσεις ε, του Συμφώνου σταθερότητα και ανάπτυξη. Και όταν είδαμε ότι η Ελλάδα έχει ένα υπερβολικό χρέος, θελήσαμε επίσης να δούμε ποιε ήταν οι χώρες αυτές οι οποίες δεν είχαν λάβει καμία προειδοποίηση και που είχαν δανειστεί τεράστια ποσά πέρα από την Ελλάδα και είδαμε ότι αυτό ίσχυε για πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά αυτόν τον τρόπο διατρέχαμε πολύ σημαντικούς κινδύνους. Και ξέρετε ότι ε, εξάγαμε επίσης πάρα πολύ προς την ε, Ελλάδα. Θα έπρεπε να είχαμε συμβάλει περισσότερο. Συντοπίσαμε ότι θα έπρεπε να υπήρχε ένα υψηλότερο επίπεδο λεγγύης Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε λοιπόν την Ελλάδα. Ορισμένοι τότε είπαν ότι θα έπρεπε να βγει από την Ευρωζώνη, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν είχαμε κάνει κάτι τέτοιο, τότε άλλοι κερδοσκοπικοί φορεί ή άλλε αγορέ θα περιμένουν, αν θέλετε, την επόμενη χώρα η οποία θα έβγαινε από την Ευρωζώνη. Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, ακόμα και η Γαλλία. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο ελεγγύη. Θα πρέπει τώρα να έχουμε και ένα σταθερό σύστημα διακυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρειάστηκε να καλύψει ουσιαστικά την έλλειψη μιας κοινή οικονομικής, δημοσιονομικής και νομισματικής διακυβέρνησης στην Ευρωζώνη. Πρέπει λοιπόν αυτό το καθεστώς διακυβέρνησης Ευρωζώνης να ενισχύσουμε και να ενθαρρύνουμε έπειτα ορισμένα κράτη-μέλη να προχωρήσουν στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους. Αναφερθήκατε επίση στην κοινωνική διάσταση, το καταγράφω και αυτό. Θα έπρεπε όντω ορισμένε χώρε, ιδίω στην Ανατολική Ευρώπη, να αυξήσουν του πιο χαμηλού μισθού του. Πρόσφατα άκουσα έναν υπεύθυνο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που μα είπε ότι, υπάρχει, ότι δεν υπάρχει αρκετό πληθωρισμό, ότι υπάρχει ένα έλλειμμα πληθωρισμού. Αν αυξάναμε του μισθού σε κάποιε χώρε Ανατολική Ευρώπη, ενδεχομένω να καταφέρναμε τελικά να αυξήσουμε τον πληθωρισμό και να φτάσουμε σε αυτό το ελάχιστο επίπεδο το οποίο πρέπει να έχει προκειμένου να μπορούν να λειτουργούν εύρυθμα οι οικονομίες μας. Θα μπορούσαμε και αυτό λοιπόν να το αναφέρουμε σε αυτή την έκθεση. Τώρα, για τις τροπολογίες σας θα πρέπει να τις καταθέσετε μέχρι τις 8 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα το αργότερο και εφόσον ο κύριος Γκάιερ ήρθε στη συνεδρίασή μας θα ήθελα να του δώσω ευθύ αμέσω το λόγο για να μας μιλήσει για τις αιτήσει μεταφοράς στα πλαίσια του προπολογισμού του 2017. Ίσως να ακούσουμε όμως πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Ρέλα, για να δούμε τι έγινε με αυτά τα αυτόνομα εμβάσματα τα οποία δεν περνάνε βέβαια από την Επιτροπή Προπολογισμού τη δικιά μας, για τα οποία βέβαια υπάρχει ένα πολύ σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο και για τα οποία όμως θα πρέπει εμείς να ενημερωθούμε. Έχει το λόγο λοιπόν εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να μοιραστώ με τα μέλη της Επιτροπής τρία ενημερωτικά σημεία. Πρώτα απ' όλα, όπως είπε και ο Πρόεδρος, πληροφορίες για τις μεταβιβάσεις. Ε, επίσης να αναφερθώ στο που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά για την αποδέσμευση κονδυλίων και τρίτον ε, η υλοποίηση του προπλησμού του 2017 ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, το κεφάλαιο 1β δηλαδή τη συνοχή πρώτα ή μεταβιβάσεις σε ό,τι αφορά τις, δημοσιονομική αρχή τι σχετικέ μεταβιβάσει είναι ενημερωμένη η Επιτροπή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκάιερ για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Ορισμένε φορέ οι προτάσει που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν επίγουσε και πραγματικά εκτιμήσαμε το γεγονό ότι και αυτό αλλά και ο πρόεδρο συμφώνησαν να τεθούν στη ψηφοφορία γρήγορα. Επίσης να σας πω ότι όπως κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρχή του Ιανουαρίου θα παρουσιάσει τις μεταφορές, τις μεταβιβάσεις ε, του τέλους του έτους, όπως τα, αναφέρουμε. Είναι μια μεταβίβαση στα πλαίσια του άρθρου 197 του οικονομικού κανονισμού, βάσει του οποίου μεταβιβάζουμε ε, πληρωμές από όλο τον προπολογισμό προς τα προγράμματα που βρίσκονται υπό κοινή διαχείριση. Προς τη συνοχή δηλαδή, την ε, γεωργική ανάπτυξη, την αλληλεία, το ΆΜΙΦ, το ISF, αυτή η μεταφορά την προετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή, να μένουν πληροφορίες από τις γενικές διευθύνσεις και σκοπεύουμε να το διαβάσουμε στην Δημοσιονομική Αρχή στις 4 Ιανουαρίου. Το όριο που προλέπει ο οικονομικός κανονισμός είναι η 10, η 10 Ιανουαρίου. Ε, να περάσουμε τώρα στις μεταφορές, τις μεταβιβάσεις που κάνει αυτόνομα ε, η Κομισιόν στα πλαίσια του άρθρου 26 του Οικονομικού Κανονισμού πάνω από χίλιε τέτοιου είδου μεταβιβάσει γίνονται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μεγάλη πλειοψηφία εξ αυτών σχετίζονται με κάποιε βελτιώσει σε ό,τι αφορά τις πληρωμές. Ε, είναι μια συνηθισμένη διαδικασία. Προσαρμόζουμε τις ε, πληρωμές ανάλογα με τις ανάγκες, ανάλογα με το ποια προγράμματα χρειάζονται ε, περισσότερα χρήματα και ποια λιγότερα. Από εκεί και πέρα, ένας περισσότερος αριθμός μεταφορών έχει να κάνει ε, για τις αναλήψεις, έχει να κάνει με τις αναλήψεις υποχρεώσεων. Οι πιο πολλές έχουν να κάνουν με το κεφάλαιο 3 και το κεφάλαιο 4. Στο κεφάλαιο 3 μπορώ να το συνοψίσω σε τρεις επιχειρήσεις. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια μεταφορά από την εσωτερική ασφάλεια ε, και τα σύνορα δηλαδή προς την αστυνομία, 18 εκατομμύρια, πάντα στο πλαίσιο της εσωτερικής ασφάλειας, στα πλαίσια του πακέτου καταπολέμησης τρομοκρατίας που εγκρίθηκε τον, Οκτώβριο τον Οκτώβριο φέτος. Επίσης, λόγω της καθυστερημένης έγκρισης της νομικής βάσης για το σύστημα εισόδου-εξόδου, τα κονδύλια τα οποία ήταν αρχικά να διαπανηθούν στα πλαίσια του ISF σύνορα, μεταφέρθηκαν στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν και το σύστημα πληροφοριών θεωρήσεων, το VIS δηλαδή και το SIS. Και ε, πλέον ε, δαπανήθηκαν για το 2017. Τρίτον, επειδή ο οργανισμός ΕΑΣΟ ζήτησε ε, υποστήριξη, ενίσχυση των δυνατοτήτων ε, ε των επιχειρησιακών, ιδιαίτερα στην Ιταλία και στην Ελλάδα, έχουμε μεταφέρει και 14 εκατομμύρια προς την ΕΑΣΟ από το πρόγραμμα ΑΜΙΦ. Σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο 4 τώρα, ε, υπάρχουν κάποιες ε, υποχρεώσεις τις οποίες τις μεταφέραμε προς, ε, στο ENI, στο ΕΠΑ, στη CFSP για τους εξής λόγους. Εντός του ECI η προπαρασκευή των project ε, για την Κεντρική Ασία είχαν καθυστερήσει. Τα project αυτά μπορούν να υλοποιηθούν μόλις το 2018. Έτσι λοιπόν μεταφέραμε μέρος ε, των υποχρέωσεων αυτών για να καλύψουμε πιο επίγουσες ανάγκες στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και στη Μιανμάρ. Έγινε λοιπόν η μεταφορά, η μεταβίβαση προς τις ανάλογες ε, τις σχετικές ε, ε, δημοσιονομικές γραμμές. Ό,τι αφορά το όργανο ε, σχετικά με τη γειτονία, ε, και εδώ έχουμε, έχουμε κάνει κάποιες μεταφορές λόγω προγραμμάτων που δεν εφαρμόθηκαν και κάποια χρήματα από το ENI από το μαξιλάρι ευελιξίας που μεταφέρθηκαν ε, προς την Νότια Μεσόγειο και προς την, ε, τις δημοσιονομικές γραμμές για τη μείωση της στόχιας στα πλαίσια της ανατολικής εταιρικής σχέσης, στα πλαίσια του ΕΠΑ τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μεταφέρει κάποιε υποχρεώσει από, από τις των Δυτικών Βαλκανίων, ιδιαίτερα τη Βοσνία, Ερζεγοβίνη και τη Σερβία, προ το πρόγραμμα ε, το που αφορά πολλές χώρες, ε, σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά προγράμματα στέγασης. Επίσης υπάρχουν και κάποιες αναλήψεις υποχρεώσεων που έχουν να κάνουν, που μεταφέρθηκαν από κάποιες γραμμές EPA προς τη μεσομική γραμμή, ε, όπου υπάρχουν ανάγκες σε, σε, χρηματοδότηση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία για να, συμπληρώσουμε την εικόνα από τα πλαίσια του προβλησμού για τη CFSP και την εξωτερική πολιτική δηλαδή έγιναν και εκεί κάποιες μεταφορές ό,τι αφορά υποχρεώσεις είναι ε, δύσκολο να καθορίσουμε τις ακριβείς δημοσιονομικές ανάγκες εκ των προτέρων όταν δηλαδή ε, λαμβάνει χρόνο του σχέδιο προπολογισμού, διότι σε μεγάλο βαθμό αυτές οι ανάγκες δεν μπορούν να προβλεφθούν και πρέπει να μπορούμε να προσαρμοστούμε και να μεταφερθούν οι σχετικές υποχρεώσεις ε, καθώς ε, οι ανάγκες προκύπτουν μετά από αποφάσεις του Συμβουλίου. Και να ολοκληρώσουμε το θέμα με τις μεταφορές, να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης έχει τη δυνατότητα να κάνει μια αυτόνομη μεταφορά προς την ανθρωπιστική βοήθεια ε, στο τέλος του έτους εφόσον προκύψει κάποια κρίση μετά την 1η του Δεκέμβρη. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πράξει αυτό πρέπει να ενημερώσει άμεσα το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτήν την μεταβίβαση. Έως τώρα δεν έχουμε λάβει κάποιο αίτημα από την Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ για μια τέτοια μεταβίβαση αλλά είναι κάτι το οποίο το έχουμε προβλέψει και στο προπολογισμό μας ε, υπάρχουν 22 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν για μια τέτοια μεταφορά ε, εάν και εφόσον ε, προκύψει τέτοιο αίτημα. Τα τελευταία πέντε χρόνια πάντα ε, είχαμε μια τέτοια ανάγκη το Δεκέμβριο συνήθως αφορούσε βεβαίως την κρίση στη Συρία. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ ε, σε ό,τι αφορά ε, το θέμα των decommitment τις αποδεσμεύσεις 4,7 ε, δισεκατομμύρια έχουν αποδεσμευθεί περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν τα περισσότερα ποσά αφορούν το κεφάλαιο 1β 2,9 δις και στο 1α 0,9 δις για τις λοιπές τα λοιπά κεφάλαια 2, 3 και 4 το επίπεδο αποδεσμεύσεων ε, δεν είναι ε, ασυνήθιστο. Να σας πω τώρα για το 1β και το 1α όμως. Για το 1β εδώ έως τώρα είχαμε 2,7 δισεκατομμύρια αποδεσμεύσεων ε, για τα προγραμμα 2007 2007-2013 τα μέλη θα γνωρίζουν ότι τα, οι τα κράτη-μέλη τους να υποβάλουν ε, δηλώσεις εξόδων ήταν 31η Μαρτίου φέτος, δηλώσεις δαπανών και έκτοτε έχει ξεκινήσει η διαδικασία ε, ολοκλήρωσης, κλεισίματος των προγραμμάτων αυτών. Αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί και του χρόνου του 2018 αλλά και το 2019. Έτσι λοιπόν η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των αποδεσμεύσεων σχετίζονται με το κλείσιμο ε, των προγραμμάτων της περίοδου 2007-2013. Υπάρχουν και 255 εκατομμύρια τα οποία αποδεσμεύτηκαν από τα παλιά προγράμματα για την περιοδο 2000-2006, δηλαδή, ακόμα πιο πολλές παλιές υποθέσεις. Ε, αυτά συνδέονται με κάποιες δικαστικές αποφάσεις και υπάρχουν και επίσης 400 ε, εκατομμύρια ε, που συνδέονται, που, που, όπου εκκρεμούν από περιπτώσει δικαστικέ υποθέσει που θα κρίνουν την τύχη αυτών των χρημάτων για την περίοδο 2006 πάντα. Τώρα, στο 1α είχα μια σημαντική αποδέσμευση σε ό,τι αφορά ε, τι μεταφορέ ε, στα πλαίσια του ΣΕΦ, αλλά δεν έχει να κάνει με το πρόγραμμα του ΣΕΦ, έχει να κάνει με τα, τον προκάτοχο του ΣΕΦ, δηλαδή τα προγράμματα TEN, για τα οποία η ημερομηνία υποβολής προσφυγών από τα κράτη-μέλη ήταν η 1η Ιανουαρίου φέτος, και εκεί λοιπόν έχει ξεκινήσει τώρα η διαδικασία του να κλείσουν ε, τα προγράμματα TEN-T και ως τώρα είχαμε αποδέσμευση της τάξης των 647 εκατομμύριων ευρώ στον τομέα των μεταφορών. Ε, στο 1α επίσης να πούμε ότι υπήρξαν αποδεσμεύσεις ε, και για τον ε, ε, προκάτοχο, τον πρόγονο του κόσμου, εν τα, στα προγράμματα ανταγωνιστικότητα για μικρομεσαίε επιχειρήσει, παραδείγματο χάρη, για την περίοδο 2001-2006, για την περίοδο 2007-2013. Αυτέ οι αποδεσμεύσει έχουν να κάνουν με το γεγονό ότι τα, τα παλιά οικονομικά μέσα ολοκληρώνονται ε, όταν διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος και οι όποιες δεσμεύσεις υπήρχαν τότε ε, δεν είναι πλέον απαραίτητες για να καλυφθούν κάποια, ε, κάποιες απώλειες, κάποιες, ε, κάποιες ζημιές πλέον αποδεσμεύονται εξού και τα χρήματα αυτά, το ποσό αυτό στο οποίο αναφέρθηκα. Τώρα, για την εφαρμογή του προπολογισμού, την υλοποίηση, θα αναφερθώ βεβαίως εδώ στο κεφάλαιο το οποίο αφορά περισσότερο τα δικά σας μέλη, το 1β. Τα κράτη-μέλη συνεχίζουν να υποβάλλουν ε, σε πολύ αργούς ρυθμούς τις, αιτήματα πληρωμών, πολύ πιο κάτω, όπως περιπτώσει, από τα προβλεπόμενα επίπεδα. Έως τώρα έχουμε 5,8 δις τα οποία δεν έχουν καλυφθεί ακόμα από αιτήματα κρατών μελών. Η Κομισιόν πληρώνει 90% ε, των αιτημάτων αυτών. Ε, αν λάβουμε υπόψη μας ε, τις υπάρχουσες πληρωμές αλλά και άλλες που έχουν υποβάλει τα κράτη-μέλη και δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, ακόμα πρέπει να λάβουμε ακόμα 5 δηλαδή, ε, αιτήματα πληρωμής ε, που να φτάνουν στο ποσό των 5 δισεκατομμυρίων για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην πλήρη υλοποίηση. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με τα κράτη-μέλη μας λένε ότι αυτό είναι φυσιολογικό και ότι όλα αυτά θα υποβληθούν ε, αργότερα εντός του μήνα, του Δεκέμβρη δηλαδή. Όμως ε, το μέγεθος είναι πολύ μεγάλο και υπάρχει βεβαιότητα. Η Κομισιόν θα κάνει ό,τι πανέ από το χέρι της βέβαια για να επεξεργαστεί όλες, όλα αυτά τα αιτήματα εφόσον βεβαίως τα λάβουμε εγκαίρως. Επ' αυτή τη βάση λοιπόν, παρότι εμείς συνεχίζουμε ε, να λαμβάνουμε καθυσυχαστικά μηνύματα από τα κράτη-μέλη, σήμερα εγώ δεν μπορώ να σας εξασφαλίσω ότι ο προπλεσμός που έχει ψηφιστεί στο πλαίσιο του 1β θα μπορέσει να υλοποιηθεί πλήρως. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιένς Γκάιερ τώρα έχει το λόγο, ο εισηγητής μας για τον προπολογισμό του 2017. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον ε, εκπρόσωπο της Επιτροπής για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Δεν είμαι απόλυτα βεβαίως κατά πόσον ε, τα κατέγραψα όλα σωστά, αλλά να κάνω κάποιες ερωτήσεις, ε, αν μου επιτρέπετε. Αν σωστά κατάλαβα, είπατε για τον ε, πρώτο τομέα της αυτόνομης μεταφοράς να ε, ε, γίνονται χιλιάδες, είπατε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο. Είναι ο μέσος όρος αυτός. Τι στοιχεία έχετε κάθε χρόνο στη διάθεσή σας. Δώσετε και κάποια παραδείγματα τα οποία ήταν εντυπωσιακά και από το ύψος τους και από πλευράς περιεχομένου. Και θα πρέπει να σκεφτούμε ενδεχομένω τέτοια ζητήματα. Γιατί που και που έχουμε μεταφορές, για παράδειγμα 14 εκατομμύρια από τα Μευστενεάζω, σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν υπάρχουν τέτοιες ε, διαφωνίες για μεταφορές ε, στον προπολογισμό σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μεταξύ κρατών μελών σε κάποιες περιπτώσεις. Νομίζω ότι αν υπήρχε πιο σταθερή και πιο τακτική ενημέρωση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδεχομένω να μπορούσαμε να κερδίσουμε επιχειρήματα σε ό,τι αφορά τι εκκρεμίε διαπραγματεύσει. Αυτές λοιπόν τις χίλιες αυτόνομες μεταφορές. Θα μπορούσατε να μου πείτε κάποια στοιχεία παραπάνω. Σε τι τομείς και σε τι ύψος κινούνται αυτές οι μεταφορές. Γιατί ως Επιτροπή Προϋπολογισμού δεν θέλουμε να μας ενημερώνετε προφανώς για κάθε 50.000 ευρώ. Αλλά όταν μιλάμε για εκατομμύρια, νομίζω ότι θα πρέπει να κάτσουμε να συζητήσουμε. Και αυτό φυσικά είναι θέμα δημοσιονομικής τάξης πιο πολύ, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε πότε ενημερώνεται και παρεμβαίνει η, η υπηρεσία, το σώμα χάραξης του προπολογισμού. Και νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική τάξη. για τις ενδιάμεσες, ε, τα ενδιάμεσα ποσά. Είπατε 4,7 μέσα δεσμεύσεις ε, αποδεσμεύτηκαν σε ό,τι αφορά το 2017. 2,9 δισεκατομμύρια αφορούν την κατηγορία 1β και από ό,τι κατάλαβα ότι πάνω από 100 από αυτές έχουν να κάνουν με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και όχι με την τρέχουσα. Αυτό μας φαίνεται αρκετά εύλογο. γιατί αν πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο δεν συνεχίζεται, αλλά για το οποίο έχουν δεσμευτεί μέσα, έχει νόημα να ανασταλεί. Αλλά θα ήθελα να συζητήσουμε κάποια στιγμή, όχι σήμερα, αλλά κάποια στιγμή το κατά πόσο θα μπορούσαμε να βγάλουμε συμπεράσματα από το γεγονός αυτό σε ό,τι αφορά δηλαδή την έλλειψη πόρων στην κατηγορία 1β και τα κρεμία αυτά προγράμματα τα οποία δεν συνεχίζονται. Εδώ πέρα υπάρχει κάποια ανακολουθία. Δεν ξέρω αν έχετε διάθεση να το συζητήσετε αυτό τώρα. Αυτό τι καταδεικνύει, ότι σε κάποια πρώτη προγραμματική περίοδο τα κράτη-μέλη ήταν σε θέση να δεσμεύσουν πόρους, αλλά στη συνέχεια διαπιστώνεται ότι δεν ε, συνεχίζονται τα προγράμματα και σήμερα δεν υπάρχει καν δέσμευση πόρων, γιατί οι αξιώσεις και οι όροι που τύφονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δέσμευση των μέσων είναι υπερβολικά αυστηροί και υπερβολικά υψηλοί. Αυτό βέβαια είναι από τη μία καλό σε ό,τι αφορά τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων, αλλά αυτό που δεν μπορεί να αποτελεί το στόχο μας είναι να δοσμεύονται χρήματα για προγράμματα τα οποία δεν υλοποιούνται. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει φυσικά ροή των πόρων αυτών και αν δεν είναι τα κράτη-μέλη σε θέση να χρηματοδοτούν, θα πρέπει να δούμε πώς ε, καταρτίζουν τη στρατηγική τους ε, σε τέτοια προγράμματα. Έκανα έλεγχο του προπολογισμού επί πέντε και πλέον έτη και τακτικά λοιπόν είδα έκθεση του λεκτικού συνεδρίου σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά αυτά μέσα και τα κράτη-μέλη τα οποία και μιλώ για τη Γερμανία σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη χρήση πόρων για τον λιμένα στη Γερμανία δεν ήταν ε, η αρμόζουσα. Δεν είναι λοιπόν πάντα τα κράτη-μέλη αυτά τα στοιχεία. Μετά από όλα αυτά όμως να σας πω κατά πόσον πιστεύετε ότι υπάρχει από πλευράς περιεχομένου κάποια σχέση μεταξύ των δύο αυτών γεγονότων. Και σε ό,τι αφορά τη ροή στην κατηγορία 1Β. Θα ήθελα να ρωτήσω αν σωστά κατάλαβα ότι πρόκειται για 5-8 δισεκατομμύρια από τα μέσα τα οποία το 2017 διατεθήκαν για τα περιφερειακά, τα ταμεία περιφερειακής στήριξης για τα κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα υποβάλει τους λογαριασμούς και δεν μπορούμε ακόμα να είμαστε βέβαιοι κατά πόσο όντως έχουν δαπανηθεί αυτά τα πόσα όντως. Σωστά κατάλαβα λοιπόν. Μάλιστα. Μπορείτε να απαντήσετε πολύ σύντομα στο γενικό μας συζητητή. αναφέρομαι στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ή ενδεχομένως να ακούσουμε και τους άλλους συναδέλφους τώρα και να απαντήσετε συνολικά, αλλά δεν νομίζω ότι θέλει να πάρει κανείς το λόγο, έτσι δεν είναι. Εγώ να κάνω απλώς μία παρατήρηση επί της ουσίας τη βλέπουμε. Οι αυτόνομες αυτές μεταβιβάσεις αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα τελικά της ενεργούς διακυβέρνησης ουσιαστικά των των πόρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφερθήκατε αυτή τη στιγμή σε 5 εκατομμύρια, ενώ έχουμε 14, για την έχουμε 14 εκατομμύρια με τη μορφή αυτόνομων μεταβιβάσεων. Αυτό καταλαβαίνετε ότι ε, μας εκπλήσει κατά κάποιο τρόπο. Κάθε φορά που περνάμε σε τριμερή διάλογο και προσπαθούμε εμείς να έχουμε κάποιους διακανονισμούς και κάποιες διευθετήσεις, ουσιαστικά σας εκλυπαρούμε για πολύ πιο μικρά ποσά, βλέπουμε παράλληλα ότι μέσω αυτών των αυτόνομων μεταβιβάσεων δίνεται δύο και τρει φορέ περισσότερα ποσά από αυτά που ζητά τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια των τριμερών διαλόγων. Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν μα πληγώνουν αναγκαστικά, αλλά ουσιαστικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις, τα μελλοντικά αιτήματα τα οποία θα κάνουμε ω αρμόδια του προπολογισμού αρχή. Έπειτα, όσον αφορά τον τομέα 4 και τι συνέβη εκεί. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκάιερ για τις ερωτήσεις του. Θα προσπαθήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Καταρχάς, όταν λέω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε περίπου χίλιες αυτόνομες μεταβιβάσεις και ότι αυτές κάνει σε αιτήσια βάση, αυτός είναι ένας μέσος όρος ένα χρόνο μπορούμε να έχουμε 800 τέτοιε, ένα άλλο χρόνο 1200 τέτοιε μεταβιβάσει. Πάντω κάθε χρόνο έχουμε εκατοντάδε τέτοιε αυτόνομε μεταβιβάσει. Και αυτέ λαμβάνουν χώρα και θα έλεγα ότι το 95% μεταβάσεων αυτών έχουν να κάνουν με την προσαρμογή των πιστώσεων πληρωμών. Γίνονται δηλαδή διευθετήσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου. Ξέρετε ότι έχουμε ένα προπολογισμό όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών. Έχουμε επιμέρους γραμμές του προπολογισμού. Ο δημοσιονομικός πάντως κανονισμός μας δίνει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους να προσαρμόζουμε τις πληρωμές αυτές καθώς ανακύπτουν νέες ανάγκες ή αποσαφηνίζονται οι πραγματικές ανάγκες των προγραμμάτων και προφανώς λειτουργούμε πάντα και μόνο στα πλαίσια του δημοσιονομικού κανονισμού. Όταν ανάγκες μας υπερβαίνουν το δημοσιονομικό κανονισμό τότε απευθυνόμαστε σε εσά και ζητούμε να εγκριθεί μια έκτακτη τέτοια μεταβίβαση επιστώσεων. Πάντω, εκατοντάδε τέτοιε αυτόνομε μεταβάσει προκύπτουν σε τέτοια βάση για μικρά συνήθω ποσά, τα οποία καταλήγουν όμω αθρηστικά να είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό, ακριβώ επειδή είναι πολλέ και γραμμέ του προπολογισμού επί των οποίων γίνονται τέτοιε μεταβιβάσει και επί των οποίων προκύπτουν τέτοιε ανάγκε. Αν πραγματικά τώρα χρειάζεστε πιο λεπτομερεί πληροφορίε για τι μεταβάσει αυτέ, θα μπορούσα να δω πώ μπορώ να σα δώσω αυτέ τι πληροφορίε. Εγώ φανταζόμουν, να σα πω την αλήθεια, ότι θα ενδιαφερόσασταν ίσω περισσότερο για τι πιστώσει ανάληψη υποχρεώσεων. Γι' αυτό το λόγο επικεντρώθηκα στην αρχική μου παρουσίαση σε αυτέ τι μεταβιβάσει. Όσον αφορά τώρα το παράδειγμα το οποίο έδωσε ο πρόεδρο πριν από λίγο, όσον αφορά την ΕΑΖΟ δηλαδή, και το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια του έτου δίνεται να μεταβιβάσει 14 εκατομμύρια από την Άμυφ στην ΕΑΖΟ, μετά από το αίτημα βέβαια της ίδιας ε, της υπηρεσίας του ίδιου του οργανισμού, ενώ από την άλλη είναι πολύ δύσκολο, όπως είπε ο Πρόεδρος, ε, στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου και της διαδικασίας συνδιαλλαγής να σας δώσουμε επιπλέον 5 εκατομμύρια σε τούμενες πιστώσεις, όπως έγινε κατά τη διάρκεια των τρεχουσών ε, διαπραγματεύσεων, καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για δύο διαφορετικές καταστάσεις. Στην περίπτωση της συνδιαλλαγής και των σχετικών διαπραγματεύσεων, καταλαβαίνετε ότι εκεί αναφερόμαστε σε επιπλέον πιστώσεις που έρχονται να προστεθούν στα όσα πρότεινε αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα αυτόματα περνάμε στη διαπραγματεύσεις που θα πρέπει να γίνουν και με το Συμβούλιο για να δούμε τι μπορεί να δεκτεί, τι είναι εφικτό και τι όχι. Και εν προκειμένου το συμπέρασμα ήταν ότι όσον αφορά την ΕΑΖΟ αυτά τα 5 εκατομμύρια μπορούσαν τελικά να γίνουν αποδεκτά και για το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενώ για το 2017 που είναι ακόμα το τρέχον δημοσιονομικό έτος, η κατάσταση διαφέρει, γιατί κατά τη διάρκεια του έτους βλέπουμε ουσιαστικά πώς εφαρμόζονται οι πιστώσεις υποχρεώσεων, ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες και ιδίως όσον αφορά το έτος 2017 για την άμυφα προέκυψε μια πολύ διάζουσα κατάσταση. Πολλές πιστώσεις προβλέπονταν για την αθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου. Καθότι όμως ε, συνεχίζουν διαπραγματεύσει τον κανονισμό αυτό, χωρίς να φαίνεται ότι θα μπορέσει να εγκριθεί ένας νέος κανονισμός άμεσα, οι πιστώσεις αυτές οι οποίες προβλεμόντουσαν στα πλαίσια της γραμμής άμυφη για τον προπολογισμό 2017, ξαφνικά γίνανε διαθέσιμες για άλλους στόχους. Και η DG Home χρησιμοποίησε τις πιστώσεις αυτές στα πλαίσια του προγράμματος Άμυφ για να καλύψει όμως άλλες ανάγκες. αλλά μπορέσαμε ακριβώς και για αυτό το λόγο να μεταφέρουμε ένα ποσό όχι πάρα πολύ μεγάλο, αξιοσέβαστο ποσό 14 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν χρειαζόμασταν πλέον για την αθόρυνση του κανονισμού του Δουβλίνου και τα οποία μπορούσαν πλέον να περάσουν στη γραμμή προπολογισμού της ΕΑΖΟ. Όσον αφορά τις αποδεσμεύσεις, νομίζω ότι ο κύριος Γκάιερ εδώ πέρα μας ζήτησε περαιτέρω διευκρινήσεις θα μπορούσα απλώς, για να είμαι απόλυτα σαφής, όσον αφορά την συνοχή στον τομέα 1β. Μηδέν οι αποδεσμεύσεις όσον αφορά το τρέχον πρόγραμμα. Για το πρόγραμμα 2014-2020 δηλαδή δεν έχουμε, ούτε προβλέπονται αποδεσμεύσεις. 2,9 δισεκατομμύρια αποδεσμεύσεις είχαν να κάνουν με τα προηγούμενα προγράμματα. Από τα 2,9 αυτά δισεκατομμύρια, τα 2,7 έχουν να κάνουν για το πρόγραμμα 2007-2013 και για ποιο λόγο διότι είμαστε στον πρώτο χρόνο της διαδικασίας κλεισίματος των προγραμμάτων αυτών, όπου τα κράτη-μέλη έχουν πλέον υποβάλει στην αρχή του 2017 όλα τα αιτήματα πληρωμών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται πλέον να αξιολογήσει, να εξετάσει τα αιτήματα αυτά και να καταλήξει τελικά σε ένα συμπέρασμα, αν δηλαδή είναι έγκυρα, νομότυπα αυτά τα αιτήματα πληρωμών, αν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και αν τελικά μπορούν να καλυφθούν με πιστώσεις ή αν θα πρέπει ένα ποσό να αποδεσμευτεί, πράγμα το οποίο συνέβη όπως σας είπα. Τα απομείνουν τα 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν να κάνουν με παλαιότερα προγράμματα από την περίοδο 2000 έως 2006 και οποιασδήποτε δεσμεύσεις ακόμα εκκρεμούν τα ΡΑΛ, τα υπόλοιπα προσεκαθάριση δηλαδή για τα παλιότερα αυτά προγράμματα πριν από το 2007, όλα αυτά είναι περιπτώσεις που έχουν ε, μπλοκαριστεί στα πλαίσια της δικαστικής διαδικασίας. Μέρος των προβλημάτων αυτών έχουν επιληθεί μέσω δικαστικής απόφασης και επομένως ένα ποσό πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσε να δεσμευτεί για τα προγράμματα αυτά και έχουμε ακόμα και 400 εκατομμύρια ραλ, υπόλοιπα προς εκαθάριση, τα οποία θα πρέπει να δούμε αν θα μπορέσουμε να τα αποδεσμεύσουμε στο μέλλον κάποια στιγμή ή όχι. Τώρα, η ανησυχία, η διπλή αυτή ανησυχία που εξέφρασε ο κύριος Γκάιερ, μας είπε από τη μία πλευρά, μας ρώτησε, πώς οι απαιτήσει που επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη μπορούν να καλυφθούν από αυτά, καθότι πολλές φορές είναι πολύ πολύπλοκες και δεν συμβάλλουν στην ελεύθερη ροή των κεφαλαίων, ενώ η δεύτερη ανησυχία του είχε να κάνει με το αν τελικά οι πιστώσεις πηγαίνουν πραγματικά και πέρα που θα πρέπει να πάνε στους πραγματικούς δικαιούχους. Τώρα η πρώτη ανησυχία είναι ιδιαίτερα, υψηλές, ιδιαίτερα υψηλά τα αιτήματα, οι προσδοκίες, οι απαιτήσει από τα κράτη-μέλη. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προετοιμασία του επόμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να πλουστεύσουμε τα πράγματα και να μειώσουμε την πολυπλοκότητα. Αυτό το παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς και σίγουρα θα κάνουμε σχετικές προτάσεις προκειμένου να καταφέρουμε να μειώσουμε το, τη διοικητική πολυπλοκότητα που βαρύνει τα κράτη-μέλη. Τώρα, οι πιστώσεις πηγαίνουν πραγματικά και που πρέπει να πηγαίνουν. Αυτή ήταν η δεύτερη ανησυχία που εκφράστηκε. Με αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε στα πλαίσια της τρέχουσας αυτής ανάλυσης που κάνουμε κατά το κλείσιμο των προγραμμάτων και ακριβώς η ανησυχία αυτή του κυρίου Γκάιερ είναι το βασικό μας μέλημα. Αν το πόρισμα τη ανάλυση μα είναι ότι πραγματικά οι πόροι δεν πηγαίνουν εκεί πέρα που πρέπει να πάνε, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι πιστώσει δεν εκταμιεύτηκαν με το σωστό τρόπο και το αποτέλεσμα της ανάλυσης αυτής είναι η λεγόμενη αποδέσμευση, την οποία σας ανάλυσα πριν από λίγο. Όσον αφορά τώρα την εφαρμογή, την εκτέλεση του προπολογισμού, θα ήθελα απλώς να επαναλάβω τα όσα σας είπα, ότι δηλαδή Εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετοιμάτων πληρωμών από τα κράτη-μέλη. Πρέπει να λάβουμε δηλαδή έγκυρες αιτήσει πληρωμών που να υπερβαίνουν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλο του έτου από τα κράτη-μέλη, αν πραγματικά θέλουμε να εκτελέσουμε τον τρέχοντα προπολογισμό όπω αρχικά είχε προβλεφθεί. Ελπίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο απάντησα στα ερωτήματά σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κύριε Σιγητά, έχετε παρατηρήσεις. Όχι. Συμπερασματικά λοιπόν, ε, κύριε Ρέλ, μπορούμε νομίζω ήδη ευθύς ε, εξ αρχής από, το επόμενο έτος να θεσπίσουμε μια διαδικασία για να έχουμε πιο τακτικά πιο τακτική ενημέρωση ό,τι φορά αυτές τις ε, αυτόνομες μεταβιβάσεις. Είναι χαμηλά ποσά, αλλά όταν συσσωρεύονται φτάνουν σε ένα σημαντικό ποσό και καλό είναι να μας ενημερώνετε σχετικά όχι για τα πιο χαμηλά ποσά, για τα μεγαλύτερα. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα ε, τις αποδεσμεύσεις, νομίζω ότι αυτό συνάδει, επικυρώνει την ιδέα ότι θα πρέπει να έχουμε ένα απόθεμα για τις περιπτώσεις κρίσεων που θα μπορεί να ε, τροφοδοτείται ακριβώς από αυτές τις αποδεσμεύσεις. Αυτό ε, μπορεί να αποτελέσει τροφή προσκέψη εν του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου ε, Ευχαριστώ τον κύριο ε, Ρέλ γιατί ήταν ε, πολύ ακριβής στις απαντήσεις του και τώρα να περάσουμε στην ψηφοφορία με μια μικρή καθυστέρηση βέβαια και στο συγγνώμη γι' αυτό αλλά ας ψηφίσουμε τώρα. Ε, παρακαλώ ετοιμάστε τις κάρτες σας να κάνουμε πρώτα μια δοκιμή Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία της εικονική ψηφοφορία αυτή, έτσι. Δεν έχουν ψηφίσει όλοι. 24 παρόντες, αλλά έχουν ψηφίσει λιγότεροι. Κύριε Ντεπρέ, πολύ ωραία. Πέρας της προφορίας. Λοιπόν, θα πρέπει να πάρουμε θέση για την έκθεση του κυρίου, του κυρίου ε, ε, για τον τρίλογο που μόλις ολοκληρώθηκε ίσως να μπορεί να μας πει κάτι πριν από την ψηφοφορία η συγγήτρια. Ναι, ευχαριστώ. Ξέρω ότι έχουμε καθυστερήσει κάπω, αλλά επειδή είναι ένα φάκελο που ε, το έχουμε συζητήσει επί μακρόν, ε, από την αρχή του έτου αργήσαμε 8 μήνε. Ε, η διαπραγμάτευση αυτή κράτησε 8 μήνε. Καλό είναι λοιπόν να υπενθυμίσω λίγο ποιοι είναι οι στόχοι που είχαμε θέσει και να αναφερθώ και στο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων πολύ πολύ σύντομα. Είχαμε τέσσερις σημαντικούς στόχους κατά τη διαπραγμάτευση του φακέλου. Πρώτον, οι προϋποθέσεις για τις επενδύσεις που θα γινόταν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δηλαδή να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στο θέμα των δύο φύλων ε, και ενίσχυση των σχεδίων που σχετίζονται ή που, των οποίων ηγούνται γυναίκες και βεβαίως μια παράμετρος που αφορά την κλιματική αλλαγή έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, να αυξήσει έως και 35% τα χρήματα τα οποία διαθέτει για επενδύσεις ε, σε αναπτυσσόμενες χώρες και μια τέταρτη υποπαράγραφο αυτής της μεγάλης κατηγορίας είναι ο στόχος αυτός ε, που έχει εισαχθεί μετά την ε, τροποποίηση της εξωτερικής εντολής, ε, διότι στην αρχή μιλούσαμε απλά για τα καταπολέμηση των ε, αιτιών της μετανάστευσης, για να προστατευτούμε κατά κάποιο τρόπο εμείς από αυτή τη μετανάστευση. Έτσι λοιπόν εμείς θέλησαμε να έχουμε μια πιο θετική στάση Πώ πρέπει να βοηθήσουμε αυτέ τι χώρε μέσω επενδύσεων για να αναπτυχθούν, για να μπορέσουν οι ίδιε αυτέ οι χώρε να επενδύσουν σε πιο παραγωγικούς τομεί για να δημιουργηθούν θέσεις Ε, να υπάρχει δηλαδή μια ανθεκτικότητα ε, σε ό,τι αφορά τις ε, χώρε αυτέ που μα περιτριγυρίζουν. Και νομίζω ότι για αυτού του τέσσερις στόχους Αυτού του τέσσερι στόχου του πετύχαμε στην διαπραγμάτευση. Τώρα από εκεί πέρα υπήρχε ένα θέμα που αφορούσε του δείκτε, αφορούσε τη διαφάνεια, τη λογοδοσία. Ε, κάναμε ένα βήμα προ την κατεύθυνση αυτή σε ό,τι αφορά την ε, επικοινωνία που θα έχουμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα υπάρχει περισσότερη και καλύτερη πρόσβαση στι πληροφορίε, ε, χωρί βεβαίω, ε, να θίγονται οι κανόνε περί εμπιστευτικότητα. Επίση, κάναμε ένα βήμα ακόμα σε ό,τι αφορά του δείκτε που θα χρησιμοποιούνται για να αξιολογούνται όλα αυτά τα project. Αυτά τα είχαμε πετύχει ήδη πριν, την, πριν το καλοκαίρι, επί Μαλτέζικης Προεδρίας, θέλω να ευχαριστήσω μάλιστα την, το έργο τη Μαλτέζικης Προεδρία. Εκεί όμως κάπου ε, μπλοκαριστήκαμε στο φορολογικό θέμα αφενός ε, και βεβαίως ε, το δεύτερο θέμα, το θέμα δηλαδή της δυνατότητα αύξησης των διαθέσιμων κονδυλίων για αυτή τη χρηματοδότηση. Εκεί ξέραμε ότι δεν είχαμε πολλές ελπίδες βέβαια. Είχαμε την τύχη, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο φάκελο, οι εξελίξεις στην Τουρκία ε, να οδηγήσουν και το Συμβούλιο και την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο να αλλάξουν κάπως ε, την ε, ε, προοπτική τους. Μειώνονται λοιπόν κάπως οι επενδύσεις και μειώνεται και ο κίνδυνος έκθεσης στην Τουρκία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και αυτό επέτρεψε να μπορέσουν να είναι διαθέσιμα κάποια κονδύλια τα οποία εμείς ανακατανήμαμε προς τις περιοχές εκείνες που για μας ήταν σημαντικές. Ε, ε, νότος, Ανατολή, Νότια Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Δηλαδή δεν χρησιμοποίησαμε ούτε ένα ευρώ περισσότερο από αυτά που προβλεπόταν, αλλά με τα χρήματα τα οποία ήταν αρχικώς να επενδυθούν στην Τουρκία μπορούσαμε να αυξήσουμε ε, τις επενδύσεις ε, λίγο πολύ στα ποσοστά τα οποία είχαμε προτείνει αρχικά. Και σε ό,τι αφορά το αφρολογικό σκέλος, Είχαμε προχωρήσει αρκετά με τη Μαλτέζικη Προεδρία. Βεβαίω μα έμεναν ακόμα κάποια εκρεμή ζητήματα για να φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο απαιτήσεων με αυτά που είχαμε, με τον άλλο φάκελο που είχαμε συζητήσει παράλληλα για την βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Καταφέραμε τελικά να φτάσουμε σε ένα κείμενο το οποίο ευθυγραμμίζεται απολύτω με του άλλου δύο φάκελου και είναι πολύ πιο απαιτητικό σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των project ε, και κυρίως ε, με ποιε οντότητε και με ποιους ε, μεσάζοντε συνεργαζόμαστε και σε ποιες χώρες ε, λαμβάνουν χώρα αυτέ οι επενδύσει. Οπότε έχουμε δηλαδή όσοι είναι στη μαύρη λίστα, όσοι δεν συνεργάζονται, όλε όλες οι χώρες που είναι υψηλού επικίνδυνου, ε, υψηλού κινδύνου έχουν μείνει εκτό επειδή δεν πληρούν του κανόνε περί είτε ε, τους κανόνες περί πληροφοριών κτλ. Σε γενικέ γραμμέ, λοιπόν νομίζω ότι πετύχαμε τον στόχο που είχαμε θέσει διαπραγμάτευση. όπω είπα δεν μπορούσαμε τελικά να έχουμε περισσότερα χρήματα αλλά λόγω της αποεπένδυσης στην Τουρκία μπορούσαμε να επενδύσουμε περισσότερο στι περιοχέ τι οποίε εμεί είχαμε θέσει ω προτεραιότητε ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι πρόκειται για μια συμφωνία η οποία είναι αρκετά ικανοποιητική. Ευχαρίστησα προηγουμένω τη Μαλτέζικη Προεδρία για το έργο τη. Ε, θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω και την Εσθονική Προεδρία, η οποία επίση μα επέτρεψε να ε, απεμπλακούμε από το διέξοδο. Να ευχαριστήσω και κυρίως τον κύριο Μουρεσάν, Επίση, ο οποίο έπαιξε ένα διπλό ρόλο. Ε, ήταν σκιώδης συγητή εκ μέρου του ΕΛΚ, αλλά ταυτόχρονα προείδρευσε και τους τρίλογου. Ε, συμμετείχε λοιπόν ενεργά, πολύ ενεργά στι διαπραγματεύσει. Θέλω να τον ευχαριστήσω λοιπόν όλου ιδιαίτερω, αλλά και τους υπόλοιπου σκιώδης συγητέ που πραγματικά ε, μα διευκόλυναν σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ πολύ. Merci, Σας ευχαριστώ. Να δώσω και εγώ την προσωπική μου λοιπόν άποψη και να σας ευχαριστήσω για την επιμονή σας και για να σας ευχηθώ και κάθε επιτυχία για τον τριμερή αυτό διάλογο και τον κύριο Μουρεσάν. Μάλιστα λοιπόν, να ψηφίσουμε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι. Με ονομαστική κλίση. Ψηφίζουμε. Le scrutin est clos. Πέρας. 22 ψήφοι υπέρ, 4 ψήφοι κατά. Και τώρα να ψηφίσουμε για την έκθεση του κ. Κολμέλ. J'ai indiqué que le rapport numéro 7 est reporté. Είχα πει ότι το 7 αναβάλλεται. Νομίζω ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε και το θέμα. Είναι δύο κανονισμοί. Και θα πρέπει να γίνουν δύο ψηφοφορίες.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 να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, να ξεκινήσουμε με το Ταμείο Εγγύσεων. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Le scrutin Πέρας. Όντως, 22 ψήφοι υπέρ και 4 κατά. και στη συνέχεια να ψηφίσουμε για τις ε, εξωτερικές δράσεις. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Πέρα. κλου. Πέρας. 22 ψήφοι υπέρ, 4 κατά. Για την έκθεση του κ. Κόλμελ τώρα. σε ό,τι αφορά τους υπηκόους των χωρών και τους απάτριδες και το σύστημα κεντρικού εντοπισμού. Έχουμε μια προφορική τροπολογία. Το Γιουλίζα θα διαθέτει την κατάλληλη χρηματοδότηση και όσα χρειάζονται για να ασκεί τις δραστηριότητες που αναφέρεται στο άρθρο 11. Ποιος είναι υπέρ, παρακαλώ. Υπέρ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Κύριε να έχετε κάποιο πρόβλημα. Ναι, αναρωτιέμαι επί τίνος τους ψηφίζουμε. Υπάρχει προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε για το αν δεχόμαστε την προφορική τροπολογία Νομίζω ότι αυτό συνέβη και νομίζω και στον σε εκεί το ίδιο λάθο έκανε. Οπότε θα ήθελα να ξαναψηφίσουμε γιατί δεν κατάλαβα ακριβώ το αντικείμενο τη κοινωνική ψηφοφορία. Εσύ. Ε... Το αντικείμενο είναι η προφορική τροπολογία, ναι, του κυρίου Κόλμελ. Έχει κανείς αντίρρηση για αυτή την προφορική τροπολογία. Δεν βλέπω αντίρρηση. Οπότε να ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας. Κατά. Ποιος απέχει εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ α, συγγνώμη, καταπίπτει καταπίπτει τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το 8 καταπίπτει Δεν καταπίπτει. Το 8 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, με συγχωρείτε. Η τροπολογία 3. Να ψηφίσουμε εκ νέου. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, επί του συνόλου τώρα του κειμένου όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το κείμενο με 19 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 4 αποχές. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία για την έκθεση που έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 7 και 29 έχουν αποσυρθεί, τροπολογία 30 υπέρ. Κατά αποχές, νομίζω ότι εγκρίνεται, λέει ο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 κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 39 άρχεται ψηφοφορία Πέρασε. εγκρίνεται 15 υπέρ 11 κατά Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41. Έχουμε προφορική τροπολογία της 41 του κύριου Ντεπρέ. Υπάρχει αντίρρηση στην προφορική τροπολογία. Ουδής. Επομένως ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 47 καταπίπτει. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 48, μάλλον καταπίπτει 48. Έχει αποσυρθεί 14, πάμε 49 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22 μάλλον καταπίπτει. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 και 25 από κοινού υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνονται. Το σύνολο τρώτο κειμένου με νομαστική κλίση άρχιτη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 21 υπέρ, 5 κατά, συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ας περάσουμε τώρα στις αιτήσεις μεταφοράς για τα υπόλοιπα τμήματα του προπολογισμού. Να δώσω λοιπόν το λόγο καταρχάς στον κύριο Τάραντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε πολύ σύντομα να σας ενημερώσω. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ζήτησε μία μεταφορά την οποία πιστεύω ότι θα πρέπει να εγκρίνουμε νομικής φύσης. Οι υπόλοιπε μεταφορές νομίζω ότι και αυτές θα πρέπει ουσιαστικά να εγκριθούν. Δεν θα ήθελα να ανοίξω παλιές πληγές και θα ζητούσα και από τους συναδέλφους να εγκρίνουν όλες αυτές τις αιτήσει μεταφορών. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, ήταν πολύ λακωνικός. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει αντίρρηση, θεωρούμε ότι βάσει της εφαρμογής του άρθρου 25 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, οι αιτήσει αυτές μεταφοράς μπορούν να εγκριθούν χωρίς αντίρρηση, όσον αφορά δηλαδή το EDPS και το EEAS και όσον αφορά τον Ευρωπαίο Μισολαβητή. Βέβαια, την αίτηση μεταφοράς για τον Ευρωπαίο Μισολαβητή δεν την έχετε στο φάκελό σας, γιατί ε, μας έφτασε αργότερα μετά τη δημοσίευσή της. Πάντως, οι τρεις αυτές μεταφορές θεωρούμε ότι μπορούν να εγκριθούν. Έτσι δεν είναι αν δεν υπάρχει αντίρρηση. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αντίρρηση. Θεωρώ λοιπόν ότι εγκρίνονται οι τρεις αυτές αιτήσει μεταφοράς. Τώρα, θα πρέπει να ψηφίσουμε και το έμβασμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άρθρο 25 και 46 του Δημοσιονομικού Κανονισμού. Η μεταφορά αυτή, η μεταβίβαση αυτή ουσιαστικά έχει να κάνει με συγκέντρωση εδώ πέρα ποσών που υπολείπονται. Ο κύριος Τάραντα θα μπορούσε να μας πει τι κάνουμε προκειμένου. Αναφέρεστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ναι. Λοιπόν, με απόλυτη ειλικρίνεια, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε όταν εγώ δεν ήμουνα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ουσιαστικά ξεκίνησε την προηγούμενη νομοθετική περίοδο και ξέρετε ότι εμεί έχουμε ακολουθήσει τη διαδικασία αυτή παρά την ε, αποδοκιμασία που είχαμε ακούσει από τον Πρόεδρο και από ορισμένα μέλη της Επιτροπής μας. και ουσιαστικά θα μπορούσαμε να καταργήσουμε τη διαδικασία αυτή. Θεωρώ ότι θα ήταν λάθος όμως αυτό, γιατί ε, το καλύτερο θα ήταν να ολοκληρώσουμε και να κλείσουμε τη διαδικασία αυτή, καθότι είναι μια μακροχρόνια διαδικασία που έχει απασχολήσει διάφορες συνεδριάσεις στο Λουξεμβούργο, που είναι το αγαπημένο μου κράτος βέβαια, και νομίζω ότι ε, θα έπρεπε εδώ πέρα οι συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας στο καινούριο κτίριο ΚΑΔ, Κόνραντ Αντενάουερ. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να κλείσουμε εδώ πέρα με τις εκκρεμείς αιτήσεις πληρωμών, μολονότι βέβαια πολλοί έχουν αποδοκιμάσει την όλη διαδικασία. Άρα είστε υπέρ, λέει ο πρόεδρος, είστε υπέρ, έτσι δεν είναι, να δοθούν αυτά τα επιπλέον 40 εκατομμύρια Μικρότερο βέβαια το ποσό που είχε ζητηθεί πέρυσι, έτσι δεν είναι. Να ευχαριστήσω πάντως σε κάθε περίπτωση τους υπεύθυνους στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν καταφέρει να προχωρήσουν σε μια κάποια εξοικονόμηση. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να χαιρετήσουμε εδώ πέρα την εξοικονόμηση που φαίνεται να έχει γίνει στο ετηθέν αυτό ποσό. Μπορούμε λοιπόν ηλεκτρονικά τώρα να ψηφίσουμε το αίτημα αυτό μεταφοράς 40 εκατομμύρια ευρώ 40.850.000 για το κτίριο ΚΑΝΤ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται για τις μεταφοράς 19 υπέρ, 6 κατά. Τώρα περνάμε στην κτηριακή πολιτική. Θα πρέπει να αποφανθούμε για αυτό το νέο σπίτι της Ευρώπης ε, που προβλέπεται στο Παρίσι. Ένα σχέδιο το οποίο θα χρηματοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Χολμάιερ δεν μπορεί να παραστεί σήμερα. Ο κύριος Φερνάντες θα την εγκαταστήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και μιλάμε για το νέο κτίριο για τον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Παρίσι. Νέα τοποθεσία Boulevard Μαν 51 στο Παρίσι. Ενώ τώρα είμαστε στο Σαν Σερμάν. Δεν υπάρχει μεγάλη προβολή όμως του τόπου αυτού και δεν υπάρχει και μεγάλη κυκλοφορία του κόσμου. Δεν περνάει πολλοί κόσμος ε, μπροστά από τον δρόμο αυτό. Είναι παλιό το κτίριο ε, και θα πρέπει να γίνει ανακαίνιση. Και το 2018 εκπνέει η σύμβαση μίσθωσης ε, με δυνατότητα παράτασης μέχρι το 2021 ως μεταβατική περίοδο. Μετά από έρευνα αγοράς έγινε μια shortlist, μια, ένας πρώτος κατάλογος και επισκεφτήκαμε λοιπόν ε, διάφορες δυνατότητες και τελικά ε, επιλέχθηκε το εν λόγω κτίριο το οποίο σας ανέφερα για σύμβαση εκμίστοσης 20 ετών. 3 εκατομμύρια, 3.000 συγγνώμη, 3.800 τετραγωνικά μέτρα με 50 υπαλλήλου ε, από το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, υπάρχουν πλεονεκτήματα λοιπόν για το νέο αυτοκτήριο. Καταρχάς η τοποθεσία κεντρική και με μέσα δημοσίων συγκοινωνιών περνά επίσης πολλοί κόσμου ε, και αυτό σημαίνει άρα μεγαλύτερη προβολή. Και αν συγκρίνουμε το κτίριο αυτό με τα άλλα κτίρια πρέπει να διαπιστώσουμε ότι είναι λιγότερο ακριβό από τα άλλα, από τα άλλα κτίρια. 5,8 εκατομμύρια λειτουργικό κόστος 1,8 δις το έτος. Η κυρία Όλμαϊερ λοιπόν προτείνει και υπερασπίζεται λοιπόν την αυτή εκμίσθωση του νέου αυτού κτηρίου, το οποίο και εγκρίνει και εξ ονόματος αυτής σας μιλώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φερνάντες. Ο κύριος Ντεπρέ. Μάλιστα, πρόεδρε. Να μην ε, αναφέρω το θέμα του ποσού, αλλά κάτι που με ενδιαφέρει. Για 20 χρόνια λοιπόν θα μισθώσουμε ένα κτίριο 5 ε, εκατομμύρια το χρόνο η εκμισθώση. 100 εκατομμύρια. Δεν ξέρω ποια είναι το κόστος αγοράς ε, ακινήτων στο Παρίσι, αλλά για 100 εκατομμύρια νομίζω κάτι μπορούμε να αγοράσουμε. Κάτι θα μπορούμε να αγοράσουμε για 100 εκατομμύρια στο Παρίσι. Γιατί λοιπόν, αναρωτιέμαι, επιλέγουμε το leasing και όχι μια αγορά. Ερώτηση, ειλικρινής ερώτηση είναι. Και άλλη μια ερώτηση. 20 εκατομμύρια θα δαπανίσουμε στην ιστορική διαρρύθμιση. Το οποίο είναι απαραίτητο για το τμήμα του Κοινοβουλίου, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα συμμετέχει, ε, συμμετάσχει παρά περιορισμένο περιορισμένο βαθμό. 20 εκατομμύρια λοιπόν εσωτερική διαρρύθμιση. Αυτό δεν θα δώσει μεγαλύτερη αξία στο ακίνητο. Άρα δεν καταλαβαίνω τη μεθοδολογία. Δεν λέω ότι είμαι κατά τη εκμίσθωση, τη μίσθωση. Απλά αναρωτιέμαι κατά πόσον αυτό θα φέρει τον ε, Ευρωπαίο πολίτη πιο κοντά στην ευρωπαϊκή πολιτική στη συγκεκριμένη περιοχή. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αναρωτιέμαι σε ό,τι αφορά το ποσό αυτό. 20 ε, εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα ωφελήσουν ουσιαστικά τον διοκτήτη, τα οποία θα χρησιμοποιήσει αν το πουλήσει δεν μπορώ να πω ότι κατανοώ τι κρύβεται πίσω από τη μεθοδολογία αυτή. Κατάλαβα λέει και ο πρόεδρο. Ο κ. Ζουμπίχη. Όλοι ξέρουμε ότι φυσικά τέτοια κτίρια σε μεγάλες πόλεις έχουν μεγάλη σημασία και η τοποθεσία του κτίριου αυτού μας καταδεικνύει ότι περνάνε κάθε ώρα 10.000 ε, πεζοί. Και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό για την προβολή στους πολίτες και την επαφή με τον πολίτη. Νομίζω ότι ανοίγουν καλές, ε, ανοίγει καλές ευκαιρίες. Το θέμα είναι να προωθήσουμε τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι μια τέτοια τοποθεσία πρώτης κλάσης είναι πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και νομίζω ότι ιδιαίτερα στη Γαλλία είναι σημαντικό να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία σε ό,τι αφορά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Μακρόν καταλαβαίνει τι ισχύει σε θέματα δημοκρατίας, αλλά υπάρχουν διάφορα κινήματα στην Γαλλία, ξέρετε, που δεν κατανοούν τα θέματα δημοκρατίας και γι' αυτό λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό ε, να προβάλλεται σωστά ο χώρος αυτός στο Παρίσι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Άρνοτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν θα σας προκαλέσει έκπληξη το γεγονός ότι θα είμαι αντίθετος για το project αυτό εξ αρχής. Επί της αρχής το 20 της Ευρώπης με 360 μοίρες, ε, σινεμά και οθόνε. Αυτά πληρώνουν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό θα έπρεπε να ισχύει. Και ύστερα αυτό που είπε ο κύριος ε, Ντεπρέ. Αυτό θα προσεγγίσει τον Ευρωπαίο πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε όχι, όποτε είχαμε τα λεφτά, είτε ναι, οπότε θεωρώ ότι είναι προπαγάνδα και σε ό,τι αφορά τις ε, διαρρυθμίσεις που έχουν να γίνουν. Ετησίως αναφέρεται ότι πρόκειται για το ενίκιο 5,8 εκατομμύρια το έτος, χωρίς πάρκινγκ και χωρίς ΦΠΑ. Επίσης μας δίνεται μια έκπτωση 30% η οποία όμως αντιστοιχεί κατά πάσα πιθανότητα στις αλλαγέ αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν. Άρα δεν είμαι σίγουρος ότι πρόκειται για έκπτωση πραγματικά και έτσι περνάμε στα 6,55 εκατομμύρια το έτος. Που αναφέρεται στο σημείο 14 στο τμήμα 2. στο σημείο 12 επίσης αναφέρεται χωρίς ε, ΦΠΑ και χωρίς ε, χώρους στάθμευσης, ε, χωρίς πάρκινγκ. Αυτό είναι τυπογραφικό λάθος. Επίσης, όταν μιλάμε για ενοικίες 20 ετών, Θα πρέπει να υπάρχει όμως ειδική ρήτρα σε ό,τι αφορά τέτοια εκμίσθωση 20 ετών. Θα μπορούσατε να απαντήσετε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νίλσεν. Eh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με την κριτική που άσκησε ο κύριος Δεπρέ και ο κύριος Άρνοπ. Πρόκειται για μια ακριβή, πάρα πολύ ακριβή μηχανή προπαγάνδας και οι Ευρωπαίοι πολίτες μας ξέρουν μια χαρά τι είναι η δημοκρατία. Είναι χαμένα λεφτά πεταμένα στα σκουπίδια για να συντηρήσουμε αυτή τη μηχανή προπαγάνδας. Και η ερώτηση που θέσατε με βρίσκει σύμφωνο σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ιδρικών Υπηρεσιών που έχει συνάψει σύμβαση 20 ετών και δεν μπορούμε πλέον να την ακυρώσουμε, να την καταγγείλουμε. Είμαι κατά τέτοιες προπαγάνδε από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να ενημερώσουμε τον κόσμο μέσω ιστοσελίδων, μέσω των ε, επισκεπτών που τακτικά έρχονται. Δεν χρειαζόμαστε σε κάθε πρωτεύουσα οίκους Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα κοστίζουν χρυσάφι. Αυτά τα χρήματα λοιπόν θα τα αφήσουμε στον Ευρωπαϊκό Αφρολογούμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο, ο κύριο Γκάιερ. Να ομολογήσω ότι ζήτησα το λόγο όταν είδα ότι ζήτησαν το λόγο και ο κύριος Άλισον και οι υπόλοιποι. Καταρχάς λοιπόν, να διευκρινίσω και νομίζω ότι η πλειοψηφία ε, της Επιτροπής απορρίπτει την, ε, τον όρο μηχανή προπαγάνδα. Είμαι Γερμανός και έχω ε, σπουδάσει ιστορία και ξέρω τι σημαίνει μηχανή προπαγάνδας. Κέντρο ενημέρωσης είναι. Σας παρακαλώ λοιπόν ε, μην χρησιμοποιείτε τέτοιες, ορισμού του τους οποίους γνωρίζουμε από τη γερμανική ιστορία, από το παρελθόν το ιδιαίτερο. Έχουμε κατά δεύτερον μια τέτοια οργάνωση ένα τέτοιο κτίριο στην, στο Βερολίνο, στην ε, οδό Ούντερ Λίντεν. Πολύ ξεχωριστή τοποθεσία, όπως και στο Παρίσι. Απέχει αυτό πάρα πολύ λίγο από τον Brandenburg Toren, από την, ε, από την Βουλή. Και ο κύριος Ρούμπιχ έχει δίκιο όταν αναφέρεται τη συχνότητα των ε, περαστικών ε, στην τοποθεσία αυτή στο Unter Linden και πόσο ωφελεί αυτό την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα λοιπόν που ανακύπτει στο σημείο αυτό είναι το εξή. Η προώθηση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και αυτή τη εγκύτητα με τον πολίτη μετράει για, για μα. Εσεί, μάλλον όχι, δεν πιστεύετε ότι είναι έτσι. Αλλά δεν είσαστε στην ε, πλειοψηφία, να ξέρετε. Κύριε Δεπρέ, πρόεδρε. Για να μην υπάρχει σύγχυση, εγώ δεν μιλάω για τη σημασία ενό κέντρου ενημέρωση και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ αυτό που αναρωτιέμαι, κατά πόσον στέκει ο ίδιο μηχανισμό ε, και μήπω ήταν πιο ενδιαφέρον να γίνει αγοραπολισία. Και μήπω έτσι παράλληλα αυτή η, αγορα, αυτή η εκμίσθωση ουσιαστικά ωφέλει τον ιδιοκτήτη. Ερωτώ όμως το εξή από τη δικαστική άποψη. Η Επιτροπή μας είναι καθελή αρμόδια σε ό,τι αφορά την απόκτηση αυτού του ακινήτου, γιατί στο σημείωμα το οποίο λάβαμε από τον κύριο Ταζάνη, το Γιάννη, το Προεδρείο έχει ήδη υπογράψει τη σύμβαση εκμίσθωσης και άρα ίσως όλη η συζήτηση είναι ακαδημαϊκής φύσεως. Όχι, λέει ο Πρόεδρος, δεν είναι ακαδημαϊκή αυτή η συζήτηση, γιατί αν είμαστε αντίθετοι στην ε, εκμίσθωση αυτή, στην μίσθωση αυτή, θεωρώ ότι θα ακυρωθεί η δικασία και θα ξαναξεκινήσουμε από το μηδέν. Ευχαριστώ, κύριε Μάνκα. Ako kvestor e, e, ευχαριστώ πολύ. Τέτοια κέντρα ενημέρωση υπάρχουν σε πολλά κράτη-μέλη. Από άποψη σε λειτουργικότητα δεν έχει να κάνει αυτό με το κτίριο. Για παράδειγμα, βλέποντα τι γίνεται στη Ρώμη, με τα γραφεία στη Ρώμη. η σύμβαση είναι για 45 χρόνια, δεν είναι σε θέση που προβάλλεται ιδιαίτερος, προεξέχουσα, δεν είναι πολύ υπεραστική. Δεν χρησιμοποιείται για διασκέψεις ε, η ασφάλεια δε κάποιων ε, παραμέτρων δεν ε, είναι εγγυημένη. Και γι' αυτό λοιπόν θέσαμε κάποιες τέτοιες παραμέτρους για το μέλλον, για μελλοντικά για μελλοντικέ εκμιστώσεις. Και παράδειγμα, το πόσο πρέστικοι περνάνε αποτελεί μία παράμετρο. Και εδώ το σημείο αυτό στο Παρίσι είναι πάρα πολύ καλό και ευνοϊκό. 18.000 ε, πραστική ανά ε, ώρα. Και Στο Βερολίνο τα πράγματα είναι λίγο πιο χαμηλά, ε, σε ό,τι αφορά του επισκέπτε για παράδειγμα, αλλά αυτέ είναι παράμετρα που ισχύουν, που έχουμε συμφωνήσει. Έχουμε εξετάσει 50 σχετικέ τοποθεσίε και πραγματικά πρέπει να σα πω ότι εξέτασα κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Συγκρίναμε όλες τις παραμέτρους. Το γεγονός ε, ότι η τιμή είναι υψηλή ε και εγώ είμαι επί τη αρχή κατά ακριβών τέτοιων ε, project, αλλά θεωρούμε ότι πραγματικά αποτέλεσαν την καλύτερη λύση για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και παρακαλέσαμε και την γαλλική κυβέρνηση για να νοικιάσει ένα τσμήμα του κτηρίου σε περίπτωση που δεν θα χρειαστούμε όλο, όλη την έκταση για τη μείωση του κόστους. Σε άλλες χώρες θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κινητέ μονάδες ενδεχομένω για κάποιο χρονικό διάστημα, δύο-τρει εβδομάδε, όπου τα παιδιά, για παράδειγμα, από τα γειτονικά σχολεία θα μπορούσαν να επισκεφτούν το Παρλαμετάριο σε κάθε πόλη αλλά σε μεγαλούπολεις όπως το Βερολίνο, όπως το Παρίσι, είναι σημαντικό να υπάρχουν ε, τέτοιες, ε, τέτοια ιδρύματα. Μόνιμα. Αυτό εξαρτάται φυσικά από το κατά πόσο θα συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το έργο λοιπόν θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό και σίγουρα θα έχει θετική επίδραση στην αντίληψη του κόσμου και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν και έλαβε και ψήφισε το Προεδρείο υπέρ τη αποφάση αυτή. Ευχαριστώ κύριο Έλισεν, έχει τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Άκουσα τον κύριο Γκάιερ και θα πρέπει να σας πω ότι έχω να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον που έχει σπουδάσει ιστορία, ε, αλλά τμήμα της ιστορίας είναι να έχουμε και σεβασμό για την άποψη των άλλων. Και όταν λέει ο κύριος Γκάιερ ότι είναι στην πλειοψηφία και ότι η δική μου γνώμη δεν μετράει, θεωρώ ότι αυτό καταπατάει την ελευθερία έκφρασης και είναι πραγματικά ιδιαίτερα αρνητικό το ότι ο κύριος Γκάιερ ότι θεωρεί ότι δεν γνωρίζω την ευρωπαϊκή ιστορία. Να σας πω ότι και εγώ την έζησα την ιστορία αυτή και αν χρησιμοποιείτε τον όρο ναζί, ναζί ε, δεν το δέχομαι και να πλύνετε το στόμα σας παρακαλώ. Πρόκειται για τη δική μας άποψη. Ε, πιστεύουμε ότι είναι όντως μηχανισμός προπαγάνδας και είναι πεταμένα λεφτά και αυτή είναι η δική μας άποψη και θα πρέπει να μπορούμε να τη λέμε. Ναι, ακούστε, αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά ότι αυτοί που έχουν ως στόχο ε, να παρνηθούμε την Ευρώπη ε, προφανώς θεωρούν ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ του γεγονότος ότι δημιουργούμε, ε, δημιουργούμε αυτό το, το νίκο ο οποίος θα αναφέρεται στο τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λογικό μου φαίνεται. Τώρα για προπαγάνδα δεν μπορούμε να μιλάμε όμως, γιατί όπως είπε και ο Γιάννης Γκέιερ, αυτή η λέξη οδηγεί σε ατυχείς συγκρίσεις και συγχύσεις. Ο κύριος Ταράν έχει το λόγο. Ναι, επειδή γίνει λόγος για προπαγάνδα, είμαι υποχρεωμένο να υπενθυμίσω στην Επιτροπή αυτή ότι στη Γερμανία χρησιμοποιήθηκε μια πολύ πιο μικρή περίοδο από τη Σοβιετική Ένωση που κατέλαβε μέρος της Ευρώπης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Προτιμώ λοιπόν να έχουμε ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών, ευρωπαϊκά γραφεία, όχι σε κάποιο ε, προάστιο, αλλά στο κέντρο της πόλης, κοντά στο Bundestag στη Γερμανία. Θα ήθελα να θαρρύνω όμως τους συναδέλφους να αναλύσουν, ίσως ε, μετά τα Χριστούγεννα, ότι πέρα από τα κτίρια υπάρχουν και αυτοί που θα εργάζονται εκεί και που θα πρέπει να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να διανύμουν, να διαδώσουν ε, τις ιδέες της ευρωπαϊκές, να ενημερώσουν και τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Θα πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να κάνουν περισσότερα, διότι τα κτίρια, το κτίριο είναι βεβαίω μια προϋπόθεση, αλλά δεν αρκεί. Évidemment. Évidemment, mais vous... Ναι, βεβαίως. Ε, ελάτε κι εσείς ε, κύριε Ταρόν να κάνετε ε, ομιλίες εκεί. Ο κύριος Έλισεν. Πρόεδρε, Δυστυχώς εδώ στο Κοινοβούλιο μιλάμε 28 χώρες και εγώ θα ήμουν υπέρ μίας ε, γλώσσας για να μην υπάρχουν προβλήματα στη μετάφραση γιατί η λέξη προπαγάνδα είναι η κανονική λέξη στην, στα Ολλανδικά. Μπορεί να το αντιλαμβάνουν διαφορετικά ε, άλλοι άνθρωποι και να υπάρχει σύνδεση με το ναζιστικό παρελθόν αλλά εγώ πραγματικά προστασιοποιούμε. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη ε, μηχανισμός διαφήμισης αλλά έτσι έχει η Ολλανδική γλώσσα και θα ήθελα να σας πω ότι αποστασιοποιούμεθα από την ακραία δεξιά και από τέτοιες λανθασμένες ε, ε, σύνδεσεις και αποχρώσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να σεβόμαστε το ένα από τον άλλον και δεν μπορούν να θεωρείται ότι άτομα τα οποία ασκούν κριτική και βρίσκονται στην μειοψηφία να θεωρείτε ότι έχουν ε, ιδέες παρόμοιες με αυτά τα οποία υπονοήσατε. Γι' αυτό λοιπόν εγώ αποστασιοποιούμε και πραγματικά πρέπει να υπάρχει και πρόβλημα μετάφρασης. Πολύ ωραία. Σημειώσαμε αυτές τις διευκρινήσεις σας. Δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να κάνουμε εδώ δίκες προθέσεων. Νομίζω μπορούμε να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 5 κατά, 3 αποχές. Η Μόνικα Ονμάιερ θα μας προσφέρει το, το επόμενο θέμα κανονικά για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την υπηρεσία εξωτερική δράση, αλλά το έχουμε αναβάλει για την επόμενη συνεδρία στις 24 και 24 Ιανουαρίου. Υπάρχει κάτι που θέλετε να προσθέσετε εσείς υπό τα διάφορα. Μάλλον όχι. Να σας πω λοιπόν ότι η επόμενη συνάντηση θα γίνει 24-25 Ιανουαρίου. Είναι τελευταία μας συνάντηση για φέτος ως ε, Δημοσιονομική Επιτροπή. Έτσι λοιπόν σε όσους δεν ξαναδώ, καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές. La séance est levée. Πέρας της συνεδρίασης. Je m'adresse aux coordinateurs. Nous avons une réunion de coordinateurs dans les minutes qui suivent. Σε λίγο έχουμε συνάντηση των συντονιστών. Εάν δεν έχετε αντίρρηση, καλό θα ήταν να γίνει αυτή η συνάντηση λίγο νωρίτερα. Να ξεκινήσουμε δηλαδή στις 5 και 4